Κυρίε και κύριοι, να σα καλωσορίσω στην κοινή αυτή συνεδρίαση με την Επιτροπή Πολιτισμού και η συνάδελφο ε, Σιρβια Κώστα, η οποία είναι πρόεδρο τη Επιτροπή ε, για την απασχόληση, είναι εδώ μαζί μα. Σα εύχομαι και καλή χρονιά, προεπιπτόντω. Με κάθε ευτυχία. και μια Ευρώπη η οποία θα αποτελέσει δύναμη και παράγοντα προς την ειρήνη και την σταθερότητα. Äh, Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε μια πρώτη συζήτηση για την κοινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη είπα τη εκπροσώπου για θέματα κρίσεων για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τις διεθνεί πολιτισμικέ σχέσει. 8 Ιουνίου 2016 και έχουμε μαζί μας τον κύριο Τιέκο Μαράνη και τον κύριο Σαμπιέρη οι οποίοι εργάστηκαν και κατέκτησαν αυτή την ε, ενημέρωση, αυτή την ανακοίνωση. Σας ευχαριστούμε λοιπόν. Και νομίζω ότι θα έπρεπε να μακρηγορήσω, αλλά παρόλα αυτά επιτρέψτε μου να πω το εξή. Η πολιτισμική διπλωματία αποτελεί ένα ζήτημα ιδιαίτερη σημασία, ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή και όπως είπε η κυρία Μοργκερίνη, το soft και hard power, τα ήπια και τα σκληρά μέτρα πολιτικής πάνε χέρι-χέρι. Και αυτό αποτελεί, συνεποτελεί την ευρωπαϊκή στρατηγική. Το θέμα λοιπόν είναι σε εποχές μεγάλων προκλήσεων. Το θέμα των φραγμών, των εμποδίων που εμποδίζουν και παρεμποδίζουν την ε, συνεννόηση με άλλες χώρες και άλλες ομάδες. Θα πρέπει όλες αυτές λοιπόν οι προκλήσεις να ξεπεραστούν για την κοινή ανάπτυξη σε ένα κόσμο πολυμερών ε, διεθνικών σχέσεων. και τέτοιων σχέσεων εναντατικών μεταξύ των κρατών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό της πολιτισμικής διπλωματίας και θα πρέπει να αποτελέσει καταλήτη. Και σίγουρα αυτό που εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι αποτελεί αξία μας και αξίες μας έχει μεγάλη σημασία. Είναι σημαντικό λοιπόν οι αξίες μας αυτές, οι οποίες εκφράζονται άλλωστε και στο χάρτη των Εμένων Εθνών. Να τονίσουμε ότι προέρχονται από την Ευρώπη ασφαλώς, αλλά ασφαλώς σήμερα έχουν τη σημασία τους σε όλο τον κόσμο και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει η απαραίτητη κατανόηση και θεωρώ ότι η Ευρώπη αποτελεί το κατεξοχήν παράδειγμα, γιατί είμαστε, όπω ξέρετε, ενωμένοι στην πολυμορφία μας. Αυτό είναι και το σλόγγαν. Και θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει αυτή η αλληλοκατανόηση σε ό,τι αφορά την πολυμορφία αυτή που επικρατεί και να διασφαλίζονται και συγκεκριμένε αρχέ νομίζω, και αξίε. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να ισχύει και επί του προεχομένου, αλλά και τυπικά και αυτό είναι προς το συμφέρον όλων μας. Και θα πρέπει να δούμε και ποιες είναι οι πολιτικές εξελίξεις και στα κράτη-μέλη και να υπάρχει όντως αυτή η ενότητα στην πολυμορφία και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να δούμε πώς ως Κοινοβούλιο, ως Επιτροπή, ως Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης μπορούμε να τα πετύχουμε όλα αυτά και πώς μπορούμε από τα θέματα αυτά, τα θέματα περιεχομένου να εφαρμόσουμε και κάποια ε, πρακτικά ζητήματα σε ό,τι αφορά και την, ε, το χαρακτήρα των κρατών μελών. Και πριν από 100 χρόνια η είπε ότι ο πολιτισμός των Ευρωπαϊκών Εθνών είναι κατά 4 πέμπτα ο ίδιος. Ε, η ίδια προέλευση έχει και ίδιο χαρακτήρα έχει. Χριστιανοδημοκρατικό θα μπορούσαμε να πούμε και βλέπουμε λοιπόν όλες τις ε, επιρροές ε, της ρίζας της Ευρώπης από τις οποίες ε, προκύπτει και η πολιτισμική εξέλιξη. Και η τέχνη ασφαλώς αποτελεί έκφανση των πολιτισμικών αυτών εξέλιξεων και ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να είμαστε σε θέση να γεφυρώσουμε αυτές τις ε, προκλήσεις και τα χάσματα που υπάρχουν και με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μπορέσουμε να έχουμε και μια κάποια λειτουργικότητα, να εφαρμόσουμε δηλαδή συγκεκριμένα προγράμματα. Το θέμα λοιπόν είναι πώς αυτές οι γενικές αρχές μπορούν να μεταφραστούν σε συγκεκριμένα μέτρα και η κυρία Κώστα και εγώ θα σας υποβάλουμε μια σχετική έκθεση η οποία βρίσκεται στη φάση της ε, κατάρτισης στην παρούσα φάση. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην παρούσα φάση στην κυρία Κώστα και στους συναδέλφους Μαράνη και Σαπιέρη για να κάνουν την εισαγωγή. Και από ό,τι φαίνεται και από τα ονόματα των ε, δύο εισηγητών υπάρχει η Ιταλική επιρροή εντονότατη. Quando si parla di cultura. <laughs> Nix cultura in Deutschland. Τι θα λέμε για τον πολιτισμό στη Γερμανία. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ και η κυρία Κώστα σας δίνει το λόγο. Grazie onorevole Brock anche per queste parole di introduzione che condivido. Eh, σας ευχαριστώ πολύ Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι σε αυτό το στο σενάριο που παρουσιάζουμε, ε, το πλαίσιο εντός του οποίου έχουμε αυτή την κοινή συνεδρίαση και ευχαριστώ τον ε, Πρόεδρο Μπρόκ για την φιλοξενία και οι δύο επιτροπέ μα, δεν συναντώνται για πρώτη φορά. Πριν από 1,5 περίπου χρόνο συναντηθήκαμε ακριβώ για αυτό το θέμα, όταν υποβάλαμε ε, και παρουσιάσαμε τα συμπεράσματα μια υπερασκευαστική δράση που ξεκίνησε το 2011 από την Επιτροπή Επισμού του Κοινοβουλίου και ολοκληρώθηκε τρία χρόνια μετά και αποτελεί και τη βάση τη γέννηση αυτή τη πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στα ευρωπαϊκά πολιτιστικά, ε, τους και ευχαριστούμε και την Κομισιόν για αυτή την πρωτοβουλία που συγκεντρώνει πολλές από τις συστάσεις που είχαν προκύψει από αυτήν την συνεδρίαση. Είμαι ευτυχής που μοιράζομαι με τον εισηγητή ε, Μπρόκ το ρόλο του, ε, της συνεισηγήτριας και ε, θα πρέπει έτσι να δώσουμε ένα καλό παράδειγμα υπέρβασης των σιλό, των συγκεκριμένων δηλαδή ε, και ξεχωριστών θεμάτων. Η κυρία Μογκερίνη εξάλλου το μοιράστηκε μαζί με δύο επιτρόπους και εδώ συμμετέχουν τουλάχιστον τέσσερις γενικές διευθύνσεις. Είναι μια σπουδαία και σημαντική καινοτομία γιατί δείχνει ότι ε, θα πρέπει να υπάρξουν κεντρικοί άξονες για τις πολιτικές και διπλωματικές δράσεις και για τις διεθνείς δράσεις. Είμαι επίσης πεπισμένη ότι σήμερα περισσότερο από ποτέ ε, και από πολιτιστική άποψη και από την άποψη του πολιτιστικού διαλόγου αλλά και της αναγνώρισης της αξίας των πολιτιστικών δικαιωμάτων ως θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, ότι αν αυτόν δηλαδή θα έχουμε καμία προοπτική ειρήνης, ε, ειρηνική συνύπαρξη και αυτό στηρίζουμε και μέσα στο πλαίσιο των δημοκρατικών διαδικασιών παγκοσμίω. Είναι πολύ σημαντικό ότι σε σχεδόν ταυτόχρονα γεννήθηκε αυτή η στρατηγική μαζί με την μεγάλη στρατηγική της Ευρώπης ως παγκόσμιο παίκτη. Είναι ένα νέο πλαίσιο εντό του εντάσσεται εντάστηκε αυτή η νέα προοπτική και κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να τηρηθούν να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις με βάση τις οποίες θα μπορέσουμε και θα το κάνουμε από κοινού ως να δώσουμε δηλαδή μεγαλύτερο βάθος στην προστιθέμενη αυτή αξία που αποκτά η Ευρώπη με μια πιο ισχυρή ε, πολιτική σε αυτό το πλαίσιο ώστε να δούμε ποιες εταιρικέ σχέσεις υπάρχουν ήδη, ποιες συνεργασίες υπάρχουν ήδη. Όπως έλεγε και ο συνάδελφος Μπροκ, ο συνεισηγητής Μπροκ. Βεβαίως θα πρέπει εδώ να εντάξουμε και να μην αντικαταστήσουμε τη δράση των κρατών μελών, αλλά να δώσουμε ένα πλαίσιο εντός του οποίου να έχουν περισσότερη ισχύ τα ε, υποκείμενα. Δηλαδή, θα πρέπει να θεωρήσουμε τον πολιτισμό στην τέταρτο πυλώνα της βιώσιμης ανάπτυξης. Δίπλα από την οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία έχουμε και τον πολιτισμό. Και Αυτό ε, νομίζω είναι κοινή γνώμη ε, πολλών συναδέλφων. Ε, υπάρχει δηλαδή, να υπάρχει δηλαδή μια νέα προοπτική. Θα πρέπει λοιπόν όχι μόνο να έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά να έχουμε και ανθρωπισμό κοινό και οι πνευματικοί άνθρωποι, οι καλλιτέχνε, αλλά και οι οικονομικά υποκείμενα, όπω α πούμε οι βιομηχανίες, οι δημιουργικές, οι πολιτιστικές, είναι κλάδοι που δεν τους εντάσσουμε πάντοτε, ε, δεν τους μάλλον ε, ε, στηρίζουμε και δεν του επιδεικνύουμε όπω θα έπρεπε. Έχουμε επίσης νέες ευθύνες, νέο πλαίσιο και έτσι θα πρέπει να δούμε και την ευρωπαϊκή ε, πιστοποίηση, η τυποποίηση. Έχουμε διαφορές, έχουμε κοινέ όμως αξίες και μπορούμε και σε αυτήν την περίπτωση να αποτελέσουμε το παράδειγμα για το πώς μπορούμε να συνδυάσουμε την ε, γλωσσική, την πολιτιστική πολυμορφία αλλά και κοινέ αξίε. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε όλες τι δυνατότητες για κινητικότητα, για ανταλλαγή εταιρικών σχέσεων με τρίτε χώρες και να στηρίξουμε ότι πρέπει να αναπτυχθεί φυσικά αυτή η δράση, η ανοχής, πρόληψης των συγκρούσεων, αλλά και της αντιπαράθεσης που μπορεί πολλές φορές να οφείλεται στην έλλειψη διαλόγου ανάμεσα στις χώρες. Δεν θέλω βέβαια να προτρέξω γιατί θα πρέπει να δούμε και ακούσαμε και διάφορους συνομιλητές, θα πρέπει να ακούσουμε μάλλον τους συνομιλητές, θα πρέπει να ενισχύσουμε αυτή τη διάσταση της επικοινωνίας και της διακυβέρνησης που γίνεται αλλά που ε, δεν γίνεται με αρκετά δομημένο τρόπο. Θα πρέπει ο συντονισμός να είναι εγγυημένος, να υπάρχει δηλαδή πολιετής ε, προγραμματισμός ώστε να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργαστεί με τρίτες χώρες πιο οργανωμένα, αλλά και να δοθεί σημασία στα ευρωπαϊκά δίκτυα, τα πολιτιστικά. Δημιουργική Ευρώπη, Εράσμος Μούντους, Μαρή Κιουρί, πολιτιστικές πρωτεύουσες. Όλα αυτά είναι μια κληρονομιά που θα πρέπει να χρησιμοποιήσει και να αξιοποιήσει η Ευρώπη. Να σταματήσω εδώ, να πω ότι βρισκόμαστε σε μια, στην αρχή μιας πορείας που θα κάνουμε μαζί και που θα ορίσουμε και επόμενα ραντεβού και θα δώσω αμέσως το λόγο οι δύο συνομιλητές που είναι εδώ. Διέγκο Μαράνη που είναι συντονιστή πολιτική για την πολιτιστική διπλωματία στην ε, Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και μετά στον δόκτωρο Βάλβο Σαλπιέρη που είναι τμήματάρχη ε, τμήματάρχης στην Επιτροπή στην Γενική Διεύθυνση Παιδεία και Πολιτισμό. Νομίζω πω είναι ενδιαφέρον να ακούσουμε τι δικέ σα αξιολογήσει. Έχετε 10 ε, λεπτά έκαστος και μετά θα ζητήσουμε από τους συναδέλφους, ξεκινώντας με τους συντονιστές και τους κοιόδης, να πάρουν το λόγο. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλοι εκπρόσωποι της Κομισιόν εδώ. Ναι, είναι και εδώ και η DG DEFCO. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ, ο κύριος Μαράνη. Έντυπα μέλη. Δεν θα επεκτάθω πάνω από 10 λεπτά. Θέλω να σας παρουσιάσω τις γενικές ιδέες και το πνεύμα της ε, ανακοίνωσης της Κομισιόν. Ο βέλτιστος τρόπος για να το κάνω αυτό θα ήταν να επαναλάβω τα λόγια της κυρίας Μογγερίνη στην ομιλία που έκανε στο πολιτιστικό φόρουμ πέρσι. Δεν θα πρέπει να φοβηθούμε να πούμε ότι είμαστε μια πολιτιστική υπερδύναμη. Είναι ο ανοιχτός μας χαρακτήρας που μας έχει κάνει μεγάλους. Η ελευθερία μας που έχει κάνει την, ε, τον πολιτισμό να είναι ένα σημείο αριστείας για την Ευρώπη. Έχουμε δώσει ένα παράδειγμα στον κόσμο γιατί και εμείς εμπνευστήκαμε από τον κόσμο. Ο δρόμος για το μέλλον αυτός είναι, να είμαστε ανοιχτή στον κόσμο, αλλά και υπερήφανη για την πολιτιστική κληρονομιά μας. Όπως είπατε, είναι ακριβώς αυτός ο δρόμος που θέλουμε να ακολουθήσουμε με αυτήν την ανακοίνωση και την προετοιμασία μιας πολιτιστικής στρατηγικής. Θέλουμε να ξεπεράσουμε την παραδοσιακή στρατηγική παρουσίαση των επιτευγμάτων μας στην πολιτική πολιτισμού και να έχουμε μια περισσότερο εστιασμένη στις επαφές μεταξύ ατόμων, μεταξύ ανθρώπων πολιτική. Επομένως δεν πρέπει να είμαστε πατερναλιστικοί και αντί να προσπαθήσουμε να πείσουμε θα πρέπει να μάθουμε και από τους άλλους και να θεωρήσουμε ότι ο πολιτισμός είναι ένα κοινό έδαφος. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τις εταιρικές σχέσεις μεταξύ των πολιτιστικών φορέων στην Ευρώπη και στις ε, χώρες εταίρες μας και επίσης να αναπτύξουμε τις ανταλλαγές, να προωθήσουμε την παιδεία και κάθε μορφής εκπαίδευση και κατάρτιση. Γιατί θέλουμε να κατανοήσουμε την κουλτούρα με ευρία έννοια και αυτό σημαίνει τις δημιουργικές, τους δημιουργικούς τομείς, την κουλτούρα σαν μοχλό ανάπτυξης, την παιδεία και τις εκπαιδευτικές ανταλλαγές. Αυτό λοιπόν το οποίο χρειάζεται είναι να προχωρήσουμε σε μια πιο συνεργατική αντιμετώπιση, ένα πιο συνεργατικό και συλλογικό παράδειγμα. Ο κεντρικός ρόλος εδώ θα διαδραματιστεί από τα κράτη-μέλη με τα εθνικά τους πολιτιστικά ε, Ινστιτούτα. Θα είναι οι συνομιλητές μας και θέλουμε να εμπλακούν σε εγχειρήματα συνεργασίας με τις ε, εταίρες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές είναι οι γενικές γραμμές λοιπόν της στρατηγικής μας και οι συναδελφοί μου μπορούν να προχωρήσουν περισσότερο σε λεπτομέρειες σε σχέση με τα θέματα της εκπαίδευσης και της ε, ανάπτυξης που έλκονται από την κουλτούρα. Ένα τελευταίο στοιχείο ίσως, το οποίο μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα το πνεύμα της ανακοίνωσης, είναι το ότι εμείς ήδη ως Ευρωπαϊκή Ένωση πράττουμε πολλά στον πολιτιστικό τομέα. Πολλά από τα προγράμματά μας έχουν ένα πολιτιστικό περιεχόμενο. Γιατί πολλές φορές δεν ξέρουμε τι υπηρεσίες, τι κάνει μια υπηρεσία μάλλον και τι κάνουν οι άλλες. Δεν υπάρχει επαφή και συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών. Αυτή η ανακοίνωση έχει σαν στόχο να διορθώσει και αυτή την κατάσταση περαιτέρω. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ σύντομα, ωραία. Και τώρα ο κύριος Ντανκέρη. Σας ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσω να είμαι τόσο σύντομος όσο ο Διέγο. Να επανέλθω σε αυτό που είπε η κυρία Κώστα. Υπενθύμησε ότι στην ανακοίνωση αυτή έχουμε βασιστεί σε ένα μεγάλο έργο προπαρασκευαστικό που έχει γίνει εν μέρη και μαζί με το Κοινοβούλιο, με την Επιτροπή ΚΑΛΤ και με την Επιτροπή ΑΦΕΤ και φυσικά και με τα κράτη-μέλη, αλλά έχουμε και πολύ συσσωρευμένη εμπειρία μαζί με τους εταίρους μας στην εφαρμογή προγραμμάτων πολιτιστικού χαρακτήρα. Και τέλος, έχουμε και την εμπειρία που έχουμε συσσωρεύσει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χάρη στη συνεργασία που έχουμε καταφέρει να επιτύχουμε με την ανοιχτή μέθοδο συνεργασίας και προγράμματα όπως η Δημιουργική Ευρώπη. Ποιο ήταν ο στόχος όλου αυτού του παρασκευαστικού έργου, να κατανοήσουμε καλύτερα τι μπορεί να κάνει ο πολιτισμός σε διάφορους τομείς. Όλοι ξέρουμε ότι είναι αφεαυτής μια αξία η κουλτούρα, αλλά ξέρουμε μπορεί να είναι και ένας μόχλος για κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη, για συμφιλίωση των λαών, για ανάπτυξη κτλ. Έχουμε μια μεγάλη εμπειρία για τα θέματα αυτά στην Ευρώπη. Και ποιο μπορεί να είναι ο ειδικό ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο να προωθήσει τα πολιτιστικά θέματα, όπω είπε ο κύριο Μπροκ. Βασιζόμαστε στις προσπάθειε των κρατών μελών, βέβαια, γιατί ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ως Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε μια κουλτούρα από την οποία να προωθήσουμε. Αλλά ο πρώτος στόχος αυτής της, ο πρώτος πυλώνας αυτής της ανακοίνωσης είναι η πολιτιστική πολυμορφία. Γιατί κατά την άποψή μας, και να σας το πω πιο μεταφορικά αν θέλετε, βλέπουμε την κουλτούρα ως ένα χώρο όπου η δημιουργία και η ελεύθερη αλληλεπίδραση μπορούν να λειτουργήσουν. Αυτό το οποίο θέλει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να διονγκώσει αυτόν τον χώρο συνεργασίας και αυτό έχουμε κάνει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό είναι που θέλουμε να κάνουμε και σε παγκόσμιο επίπεδο για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις πολιτικές σχέσεις και να κάνουμε μια καλύτερη συμβολή στις εξωτερικές μας σχέσεις. Γι' αυτό θεωρήσαμε ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε με μερικέ βασικέ αρχέ και μία από αυτέ είναι η πρόθεση της πολιτιστικής πολυμορφίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όπως είπε και η κυρία Κώστα, σημαίνει ότι θα πρέπει να βασιστούμε σε αυτόν τον κοινό ουμανισμό με τον οποίο μπορούμε να ενισχύσουμε τις πολιτικές οι οποίες υποστηρίζουν αυτό το κοινό κληροδότημα. Όπως ο υποδιέγκο δεν είναι να προωθήσουμε και τη δική μας κουλτούρα και να αυτό επιχαίρουμε, αλλά για να βοηθήσουμε και τους άλλους να κάνουν αυτά τα οποία πρέπει να κάνουν, τους πολιτιστικούς φορείς, οι οποίοι είναι πολύ καλύτεροι από εμάς. Και υπάρχει και επίσης και ανάγκη συμπληρωματικότητας και επικουρικότητας. Θα συνεργαστούμε με τις κυβερνήσεις, με τους εμπλεκόμενους φορείς, θέλουμε να σεβαστούμε πλήρως την αρχή της επικουρικότητας. Επιπλέον και για το λόγο ότι μόνο τα κράτη-μέλη μπορούν να κάνουν πραγματικά το έργο το οποίο χρειάζεται να γίνει. Μόνο οι πολιτιστικοί φορείς σε εθνικό επίπεδο μπορούν να το επιτύχουν αυτό. Παρουσιάσαμε λοιπόν αυτήν την ε, σειρά δράσεων στην ανακοίνωση που θέλουμε να διοργανώσουμε. Θα μπορούσε να είναι διαφορετική επιλογή των δράσεων αυτών, αλλά θελήσαμε να δώσουμε έμφαση στην συμβολή της κουλτούρας στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη, όπως είπε η κυρία Κώστα, είναι βασικό στοιχείο της αηφόρου ανάπτυξης και είναι απαραίτητο να βοηθήσουμε και τους εταίρους μας να αναπτύξουν το δικό τους δρόμο προς την αηφόρο ανάπτυξη. Και επίσης είναι σημαντική η συμβολή στον διάλογο και την συμφιλίωση της κουλτούρας για να υπάρξει μεγαλύτερη και κοινωνική συνοχή. Έχουμε δυστυχώς και στην Ευρώπη αρνητικά παραδείγματα. Θυμηθήκαμε, μπορούμε να θυμηθούμε τι έγινε σε περιπτώσει όπως της Ιουκοσλαβίας, της Ιλλανδίας, της Κύπρου, ώστε η κουλτούρα να προωθήσει την συμφιλίωση μεταξύ αντιμαχωμένων πλευρών. Και ένα τρίτο στοιχείο που θέλουμε να τονίσουμε είναι η πολιτιστική κληρονομιά. Όλοι έχουμε υπερηφάνεια για την τι πολιτιστικέ μα ρίζε. και είναι απαραίτητο να μπορούμε να έχουμε ένα διάλογο για τα θέματα αυτά, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κάτι μελέτη συσσωρεύσει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Είναι χώρο χώρο όπου μπορούμε να έχουμε ανταλλαγέ απόψε με του εταίρου μα προ το κοινό συμφέρον και έχουν γίνει ήδη συγκεκριμένε δράσει προ την κατεύθυνση αυτή. Θεωρήσαμε λοιπόν να έχουμε ένα τέτοιο πανόραμα για τις συνολικές μας δράσεις, γιατί με τον τρόπο αυτό φαίνεται καλύτερα τι μπορεί να κάνει η κουλτούρα για, τα, για τους στόχους μας και επίσης δείχνει το εύρος τη παρέμβαση που θέλει να κάνει η Κομισιόν. Η ανακοίνωση αυτή παρουσιάστηκε τον Ιούνιο και από τότε έχουμε αρχίσει να εφαρμόζουμε κάποιε δράσει. Και φυσικά, αν έχετε κάποια ερωτήματα για αυτέ τι δράσει, είμαι στη διάθεσή σα. Το τελευταίο κεφάλαιο που θέλω να αναφέρω και το ίσω το πιο σημαντικό είναι αυτό των εταιρικών σχέσεων. Η στρατηγική αυτή μπορεί μόνο από κοινού να επιτευχθεί με δράση μόνο της Κομισιόν δεν μπορούμε να επιτύχουμε τα αποτελέσματα ούτε σε επίπεδο προγραμμάτων και σχεδίων, αλλά ούτε και σε συνολικό επίπεδο. Γι' αυτό, όπω είπε και ο Διέγκο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε την ενεργή συμμετοχή των Εθνικών Πολιτιστικών Ινστιτούτων και Φορέων, γιατί έχουν τη δυνατότητα να παίξουν ένα πολλαπλασιαστικό ρόλο στις δράσεις μας και να έχουν και ευρύτερη πρόσβαση σε όλους τους πόρους που υπάρχουν στα κρατη και να επιτύχουμε με αυτόν τον τρόπο ένα μεγαλύτερο αποτελέσμα. Η συμπληρωματικότητα λοιπόν μεταξύ χωρών και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να εξασφαλίσουμε ότι και η δράση αυτή θα είναι όσο δυνατόν πιο κοντά στους πολίτες και γι' αυτό οι πολιτιστικοί φορείς και εμπλεκόμενοι είναι οι απαραίτητοι εταίροι και οι δρόντες για να μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Γι' αυτό λοιπόν Έχουμε δημιουργήσει τις πλατφόρμες πολιτιστικής δράσης που δίνουν κατάρτιση, παροχή συμβουλών και είναι και ένα εργαλείο που μας επιτρέψει να, επιτρέπει να συλλέξουμε τις βέλτιστες πρακτικές. Είναι ένα εργαλείο το οποίο θα μας επιτρέψει να κατανοήσουμε και τη θέληση της κοινωνίας των πολιτών και να συνεργαστούμε καλύτερα μαζί τους. Και εκεί παίζει σημαντικό ρόλο παίζουν σημαντικό ρόλο για αντιπροσωπείε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ο στόχο είναι να γίνονται επιτοπίωση οι δράσεις σε κάθε χώρα που εμπλέκεται και οι αντιπροσωπείε της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να βοηθήσουν τη δημιουργία αυτής τη πλατφόρμας όπου θα συναθρίζονται οι τοπικοί παράγοντε στον πολιτιστικό τομέα, οι εθνικέ κυβερνήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε ήδη επιτύχει να εδραιώσουμε μερικά σημαντικά αποτελέσματα στον τομέα αυτό και θα δώσω τώρα στη συνάδελφό μου το λόγο, εάν μου επιτρέπετε, για να παρουσιάσει τη συνέχεια. Ο πολιτισμός λοιπόν πάντα ήταν τμήμα της πολιτισμικής συνεργασίας και να σας πω και ποια είναι τα πιο επιτυχή παραδείγματα από την υποστηρίξη που έχουμε παράσχει στα σε βάθος χρόνου και βάσει των τριών πυλώνων που ανέφερε ο Βάλτερ, ε, την οικονομική ανάπτυξη, πολιτισμικός διάλογος για ειρηνικές ε, σχέσεις και πολιτισμική κληρονομία. Καταρχάς, λοιπόν, σε ό,τι αφορά τον πρώτο πυλώνα, σε ό,τι αφορά τις κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις και τη σχέση τους με τον πολιτισμό. Έχουμε συγχρηματοδοτήσει την παραγωγή ενός ε, φιλμ, ταινίας που ονομάζεται Ραν, στην Ακτή Λεφαντεστού, που ε, κάνει μια αναδρομή στο στρατιωτικό ιστορικό παρελθόν της χώρας και αυτό όχι, όχι μόνο έπαιξε ρόλο στην συμφιλίωση, αλλά έδωσε και μια όθηση στον γενικό κλάδο της παραγωγής ταινιών το 2014-2015 και έκτοτε τέσσερις ακόμα ταινίες έχουν προκύψει από τη χώρα αυτή. Ε, συστήθηκε ένα σχετικό ταμείο, μια βάση δεδομένων για τεχνικούς που παρέχονται υπηρεσίες και υπήρξε κατάρτιση και τεχνικών και ηθοποιών. Σε ό,τι αφορά τον αντιπολιτισμικό διάλογο, είχαμε ένα πολύ επιτυχές project με γερμανική συγχρηματοδότηση στη Σρι Λάνκα, που επίσης συνέβαλε στη διαδικασία επανασυμφιλίωσης και προώθησε την πολιτισμικότητα και τα αποτελέσματα ήταν ε, προγράμματα ανταλλαγής για ε, πολιτισμικούς φορείς και για πανεπιστήμια. Δόθηκαν κάποιες επιχορηγήσεις για παραγωγή για κάποιες παραγωγές και κάποιες ε, τοπικές πρωτοβουλίες που είχαν τοπικό αντίκτυπο και επίσης διευκολύναμε την διοργάνωση φεστιβάλ τα οποία και αυτό με τη σειρά του συνέβαλαν σε μια επανασυμφιλίωση. Τρίτο παράδειγμα για την πολιτισμική κληρονομιά. Αυτό περιλαμβάνει τη Δυτική Αφρική και την τοπική αρχιτεκτονική. Στον Νίγηρα, για παράδειγμα, έχουμε ένα έργο όπου ε, φροντίσαμε για την διατήρηση αρχιτεκτονικής και έτσι σε ένα εθνικό μουσείο προβάλλεται η παραγωγή τέτοιων πύλινων αντικειμένων με πλήθες μια σειρά δραστηριοτήτων που προωθεί γενικώ την εθνική κληρονομιά και πάνω από 100 άτομα εκπαιδεύτηκαν και απέκτησαν την τεχνογνωσία για την ε, παραγωγή των αντικειμένων αυτών. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, λέει η κυρία Κώστα, πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα παραδείγματα και τώρα θα δώσω το λόγο στους εισηγητές, στους σκιώδους εισηγητές καταρχάς και μετά στους υπόλοιπους συναδέλφους. Ποιος θα θέλει να πάρει το λόγο, παρακαλώ. We can alternate one from Culture Committee, one from... Να ακούμε έναν συναδελφό από την Επιτροπή ΑΦΚΟ και έναν την Επιτροπή Πολιτισμού. Να αλλάξει. Χιμένες Μπαρμπάτε και μετά τον κύριο Μιλαμόν. Ε, Καλημέρα σας. Ήταν πολύ θετικό το ότι ξεκινήσαμε να μιλάμε για τα θέματα αυτά, για αυτά που είπε και η κυρία Μογκερίνη για την πολιτιστική διπλωματία και για τον πολιτισμό σε σχέση με τις διεθνείς σχέσεις. Το Κοινοβούλιο έχει ήδη εκφράσει την απόψή του στο παρελθόν με ψηφίσματα και εγώ ως εισηγήτρια για τα θέματα αυτά στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, θέλω να δείξω ορισμένα θέματα που είναι σημαντικά για μας. Είναι απαραίτητο να μπορούμε να έχουμε θετική δράση για τα πολιτιστικά ζητήματα. Παραδείγματο χάρη, θα ήθελα να αναφερθώ στα πολιτιστικά ιδρύματα που έχουμε στο εξωτερικό. Παραδείγματο χάρη το Ινστιτούτο Θερβάντες, και άλλα τέτοια πολιτιστικά ιδρύματα, τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο στο να μεταλαμβαδεύσουν τη γλώσσα, αλλά και την κουλτούρα και τον πολιτισμό, την λογοτεχνία κτλ. των χωρών μας. Και ουσιαστικά αρχίζουν να γίνονται και πολιτιστικοί πρεσβευτές της Ευρώπης, που θέλουμε όλοι να έχει ένα κοινό διάλογο, ένα κοινό λόγο, ένα λόγο ο οποίο θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ολοκλήρωση και να μπορέσουμε να μεταφέρουμε και σε άλλες χώρες την ιδέα αυτής της επιμερισμένης ε, μορφής πολιτιστικής ενότητος, ώστε και οι χώρες αυτές να μπορέσουν να αποδηθούν σε αυτό το σημαντικό εγχείρημα του να επιτύχουν αυτή την συλλογική πολιτιστική ταυτότητα. Επίσης με ενδιαφέρει πάρα πολύ η επιστημονική διπλωματία, όπως και η κουλτούρα και η επιστήμη είναι μια ήπια ισχύς, όπως λέμε, και μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ τις σχέσεις μας με χώρες εκτός της Ευρώπης. Είναι η επιστήμη αυτή η οποία μπορεί να μας συνενώσει καλύτερα, γιατί πρόκειται για θέματα τα οποία δεν εξαρτώνται από το συναισθηματικό τμήμα, από την ιστορική παράδοση, από τις παραδόσεις. Είναι ένας χώρος αντικειμενικός όπου δεν μπορούν να παρισφρήσουν, τουλάχιστον δεν θα έπρεπε να παρισφρήσουν αυτές οι υποκειμενικές απόψεις. Είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός χώρος λοιπόν και γίνονται πράγματι πάρα πολλά πράγματα προς την κατεύθυνση αυτή, ιδίως μέσα στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής Γειτονία, Όταν ήμασταν στην Τίνιδα μαζί με την κυρία Κώστα, συζητήσαμε όλα αυτά τα θέματα και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να συζητήσουμε και να προχωρήσουμε περισσότερο. Το Πανεπιστήμιο τη Τίνιδος, παραδείγματο χάρη, θα είναι τμήμα του σχεδίου Horizon 2020. Θα υπάρξει μια δυνατότητα χρηματοδότηση τη έρευνα και τη ανάπτυξη και προ το Πανεπιστήμιο αυτό. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, μπορούν να μα βοηθήσουν. Και εγώ είμαι αντιπρόεδρο στην αντιπροσωπεία του Μάγρεπ με τον τρόπο αυτό μπορούμε να αναπτύξουμε αυτέ τι σχέσει και του δεσμού με το βόρειο τμήμα τη Αφρική. Είναι περιοχέ οι οποίε μα ενδιαφέρουν ιδιαίτερα για να μπορέσουμε να εδραιώσουμε σταθερέ σχέσει και να μπορέσουμε να πραγματώσουμε κοινού στόχου με την ε, συνεργασία μας. Επίσης δεν πρέπει να παραλείψω και το πάρα πολύ σημαντικό θέμα της πολιτικής κληρονομίας, της προάσπισης ευρωπαϊκής πολιτικής κληρονομιάς. Ήμουνα πρόσφατα με ορισμένου φίλους στο Μόναχο, πέρασα από την πινακοθήκη του Μονάχου και εκεί βλέπει κανείς πόσο μεγάλο είναι αυτό το κοινό κληροδότημα που έχουμε στην Ευρώπη, στο οικαστικό αλλά και σε άλλους τομείς. Θέλουμε όμως να δούμε και τι γίνεται για τις χώρες του Μαγρέπ και της Βόρειας Αφρικής όπου εμεί θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μα, να διατηρήσουμε και το δικό του κληροδότημα, το οποίο είναι και αυτό το τμήμα τη δική μα κουλτούρα και ιστορία. Και επομένω θα πρέπει εμεί να προωθήσουμε όλα τα δυνατά μέσα, ώστε να υπάρξει προστασία και διατήρηση του τοπικού τους πολιτιστικού κληροδοτήματος προς το συμφέρον των χωρών αυτών, αλλά και για μας και για τις επερχόμενες γενιές. Αυτά είναι τα σημαντικά θέματα λοιπόν, τα οποία θα ήθελα να δείξω. Ευχαριστώ. E Σας ευχαριστώ. Και τώρα ο συνάδελφος Μίγιαν Μόνο. ευχαριστώ. Και ευχαριστώ πρώτα απ' όλα τους ε, δύο προέδρους, ε, την κυρία Κώστα και τον κύριο Μπρόκ, που συγκάλεσαν αυτήν τη συνεδρίαση. Θυμάμαι πως μα έλεγε η Σίλβια Κώστα πριν από λίγα λεπτά, ότι υπήρξε μια συνεδρίαση κοινή στην Άνοιξη του 2015, αν δεν κάνω λάθος. Εν τω μεταξύ όμως υπήρξε η ανακοίνωση της Κομισιόν εγώ πιστεύω πολύ στα όσα αναφέρονται σε, αυτό το ανακοινωθέν και ελπίζω πως έτσι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και εμείς και να βελτιώσουμε την πρόταση. Και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάποιους προβληματισμούς. Καταρχήν, ο πολιτισμός είναι ένα σημαντικό μέσο οικονομικής ανάπτυξης. Πολιτιστικός τουρισμός, για παράδειγμα, αλλά, όπως είπαμε, είναι σημαντικός ο πολιτισμός και για την ανάπτυξη ευρύτερα. Έπειτα πρέπει να τονίσουμε πως ε, ο πολιτισμός ε, είναι σημαντικός για μια ειρηνική και ανεκτική ε, κουλτούρα, νοοτροπία, διάλογος, ανοχή, αυτά να στηρίξουμε ενώ υπάρχουν άλλοι που προτάσουν τον δογματισμό και τον απολυταρχισμό. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να προσπαθήσουμε ώστε να προλάβουμε τον απολυταρχισμό και τον δογματισμό. Πρέπει δηλαδή να μπορέσουμε να προλάβουμε τη ριζοσπαστικοποίηση. Τρίτη πτυχή που ήδη έχει αναφερθεί είναι το πολιτιστική, πολιτιστική κληρονομιά. Μάλιστα αυτή η χρονιά είναι η χρονιά της πολιτιστικής κληρονομιάς. Εδώ και η Σίλβια Κώστα ήταν αυτή που στήριξε ε, την, το έτος της ε, πολιτιστικής κληρονομιάς. Συμφωνώ και επαυξάνω και γι' αυτό και υπήρξε και μεγάλη επιτυχία μετά από κάποιες πρώτες ε, αμφιβολίες. Ελπίζω πως θα είναι επιτυχής αυτή η πρωτοβουλία και να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεγάλη δύναμη σε αυτό το θέμα του πολιτισμού και πρέπει να προσπαθήσουμε εμείς να διατηρήσουμε και την πολιτιστική κληρονομιά και του υπόλοιπου κόσμου ε, σε συνεργασία με την UNESCO. Μετά από όλες τις βαρβαρότητες που έχουμε δει να διαπράττονται σε ορισμένες χώρες, ας πούμε στο Αφγανιστάν ε, πρόσφατα το τι συνέβη εκεί και το τι συμβαίνει στην Παλμύρα. Κάτι ακόμα που δεν ξέρω αν υπάρχει. μπορεί να μην, να μην το βρήκα εγώ αλλά και να υπάρχει οι ε, πολιτιστικοί δρόμοι της Ευρώπης που τη διαχειρίζεται το Συμβούλιο της Ευρώπης ε, το επόμενο χρόνο, όχι φέτος, φέτος ε, ολοκληρώνονται 30 χρόνια αυτής της πρωτοβουλίας. 33 δρόμοι, πολιτιστικοί δρόμοι της Ευρώπης που είναι πολύ σημαντικοί για να καταλάβουμε τι είναι η Ευρώπη και αυτή η πολυμορφία πολιτιστική και αλλά και ενότητα πολιτισμών που είναι η Ευρώπη. Για τους νέους μας είναι πολύ σημαντικό να μην γνωρίζουν μόνο το δρόμο του Σαντιάγο, αλλά ας πούμε την ε, Απία Οδό, τις διάφορες άλλες ρωμαϊκές οδούς. Είμαι, είμαι πεπισμένος ότι όλα αυτά θα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και δεν είναι μόνο κληρονομιά ευρωπαϊκή μα ενώνουν και με τους γείτονές μας, γιατί υπάρχουν δρόμοι που συνδέουν ας πούμε, την Ανταλουσία με το Μαγρέμπ, με το Μαρόκο. Ο δρόμος των, ε, των Σερφαδιτών, για παράδειγμα, ένα σωρό τέτοιες ε, πορείες ε, θα πρέπει να δοθεί δηλαδή σημασία σε αυτούς τους πολιτιστικούς δρόμους να χρηματοδοτηθούν. Είναι πολύ σημαντική για να καταλάβουμε την Ευρώπη και για να καταλάβουμε, όπως είπα, την Ευρωπαϊκή Ενότητα ε, που είμαστε, Ενότητα Πολιτισμών. Ενώ οι υπόλοιποι θέλουν να κατακαιρματίσουν την Ευρώπη και προτείνουν τη διάλυσή της, εμείς θα πρέπει να προτάξουμε αυτούς τους πολιτιστικούς δρόμους που μας ενώνουν. Τώρα, Εράσμο, Εράσμο Μούντι, αυτέ οι εταιρικέ σχέσεις κινητικότητα που κάνουμε με διάφορε χώρε, α πούμε με τους γειτονικέ χώρε στο Μαρόκο ή και αλλε ε, να ε, εντάξουμε και του νεου του φοιτητε που είναι το μέλλον του κόσμου, το μέλλον τη ευρωπη ε, Γι' αυτό οι, οι ανταλλαγές φοιτητών είναι πολύ σημαντικοί Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ και επειδή μας θυμήσατε το σημαντικό ραντεβού του 2018. Julie Ward, από την Επιτροπή ε, Πολιτισμού. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ όλους και νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ ευπρόσδεκτη συζήτηση αυτή που κάνουμε και πολύ χάρηκα που η υπατή εκπρόσωπο έκανε την ανακοίνωση αυτή στο ε, Φόρουμ Πολιτισμού την προηγούμενη χρονιά και νομίζω ότι πραγματικά ε, αλήθεια Εμεί που εργαζόμαστε στο τομέα του πολιτισμού καταλαβαίνουμε και κατανοούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό το πόσο σημαντικό ρόλο παίζει ω γέφυρα μεταξύ των ανθρώπων. Συχνά όταν όλα τα άλλα έχουν αποτύχει, οι πολιτισμικέ δραστηριότητε και ο διαπολιτισμικό διάλογο μεταξύ των λαών καταφέρνουν να πετύχουν τη συνέχιση σχέσεων. Και αυτό συμβαίνει ακόμα και όταν ο κόσμο δεν μιλάει καν την ίδια γλώσσα. Γιατί ο πολιτισμό συχνά μεταφράζονται σε δράσεις, σε ενέργειες. Δεν είναι μόνο αυτά που λέμε, δεν είναι μόνο λόγια. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερος που άκουσα να περιγράφεται ως χώρος ο πολιτισμός. Η συμπερίληψη λοιπόν της αρχιτεκτονικής είναι πάρα πολύ σημαντική η αρχιτεκτονική έχει πολύ σημαντικό ρόλο. Δεν είναι μόνο τα κτίρια που φτιάχνουμε, αλλά και ο χώρος που δημιουργούμε για να, ε, έρθει κοντά, να έρθουν κοντά οι άνθρωποι ή για τα φράγματα τα οποία και τα εμπόδια τα οποία ε, καταφέρνουμε να απαλείψουμε μεταξύ των ανθρώπων. Και να σας πω ότι με ενδιαφέρει ιδιαίτερως μία έκθεση για την περιφερειακή ανάπτυξη για τις περιθωριοποιημένες κοινωνίες. Και κοινότητες. Θέλαμε να προσκαλέσουμε λοιπόν εμπειρογνώμονες, αρχιτέκτονες, γιατί ακριβώς δραστηριοποιούνται στο δημόσιο χώρο και δημόσιος χώρος είναι κάτι το οποίο πολύ φοβόμαστε σήμερα. Θα πρέπει όμως να το κάνουμε δικό μας, το δημόσιο χώρο. Και υπάρχει λοιπόν μια ομάδα η οποία εξετάζει τα δημόσια αγαθά και τους δημόσιους χώρους. Τα κοινά λοιπόν είναι ένα ζήτημα και αυτό με τη σειρά του μας οδηγεί σε σκέψεις και ιδέες που αφορούν την ίδια τη δημοκρατία. Άρα θεωρώ ότι αυτό που συζητάμε, το να προσεγγίσουν λαοί, κοινότητες, άλλες κοινότητες, θρησκευτικές πολιτισμικές κοινότητες, ο πολιτισμός άλλωστε είναι κάτι το δυναμικό, το οποίο αλλάζει, το οποίο δεν περιορίζεται. Είναι σημαντική λοιπόν η έννοια του δημόσιου χώρου. Και να προσθέσω και δύο λόγια για την, τον κλάδο του τσιρκού και των ε, τεχνών του street art. Οι καλλιτέχνες ε, τσιρκού έχουν ε, μία μακρά παράδοση και το τσίρκο αποτελεί μία μορφή τέχνης που περιλαμβάνει και πάρα πολλούς προτεραιοποιημένους νέους. Είναι πάρα πολύ λοιπόν συναρπαστικός ως κλάδος. Το τσίρκο λοιπόν περιλαμβάνει ακόμα και άτομα με αναπηρίες. Είναι πραγματικά εξαιρετικός ε, τρόπος να έρχονται κοντά οι άνθρωποι. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ε, συναρπαστικό βιβλίο, το οποίο ονομάζεται Clowns Without Borders, ε, Clown Holy Σύνορα, για τους κλόουν και στη σχέση τους με τους πρόσφυγες. Να μην ξεχνάμε λοιπόν και αυτές τις μορφές τέχνης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Μπούχνερ. Σας ευχαριστώ. Έχω ένα σύντομο μοναχά ερώτημα. Α, θα τα πω στα γερμανικά, συγγνώμη. Ο πολιτισμός δεν βρίσκεται μοναχά στα βιβλία και στα μεγάλα πολιτιστικά κέντρα, αλλά και στην καθημερινή ζωή. Αυτό σημαίνει για μένα ότι ακόμα και τα ηλεκτρονικά μέσα, η τηλεόραση, το ραδιόφωνο μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο για τη μεταλαμβάνευση του πολιτισμού. Αυτό με οδηγεί να αναρωτιέμαι γιατί τα Euronews ε, έχουν πουληθεί και αυτή τη στιγμή ένας Αιγύπτιος επιχειρηματίας έχει πάρει το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών και οι υπόλοιπες μετοχές θα πουληθούν δεν ξέρω και εγώ πού αλλού και με αυτόν τον τρόπο υπήρξε αυτή η μετατόπιση του κέντρου. Ξέρετε ότι θα υπάρξει εκπομπή και θα σταματήσει παραδείγματος η εκπομπή στα περσικά. Αυτό για μένα έχει καταστροφικό χαρακτήρα. Αυτό για μένα είναι ένα πλήγμα για, την ευρωπαϊκή, για τη μεταλαμβάνευση ευρωπαϊκής κουλτούρας. Για αυτή την ερώτηση είμαι σίγουρος ότι θα απαντήσει, σίγουρη ότι θα απαντήσει ο συνάδελφος Μπρόκ στο τέλος, αλλά σίγουρα εμείς ε, γι' αυτό θέλαμε να έχουμε επαφή με την Κομισιόν για να καταλάβουμε καλύτερα τι εννοεί. Πέτερλε. Dragi kolegi, eh, jaz vesel, da στο τότσικο dnevnega reda na prvi letošnji seji. Ξεκινάμε αγαπητοί συνάδελφοι. Τη συζήτηση αυτή στην πρώτη συνεδρίαση τη Επιτροπή μα και αυτό έχει συμβολικό χαρακτήρα. Συζητάμε μια πάρα πολύ σημαντική στρατηγική γιατί ο πολιτισμό είναι ένα τομέα όπου έχουμε πολύ ανεκμετάλλευτο δυναμικό και μιλάω με τη δική μου σλοβενική εμπειρία. Όταν πήγα στην Ιγυρία στην ε, αποστολή εκλογικής παρακολούθησης εκεί, ήταν να υπάρχουν πολλές δυνατότητες για πολιτιστική συνεργασία. Χαίρομαι για το γεγονός ότι οι συνομιλητές μας ενδιαφερόντουσαν ιδιαίτερα για την πολιτιστική κουλτούρα της Ευρώπης και αναρωτιόντουσαν πώς καταφέραμε εμείς να συνδυάσουμε τις διαφορετικές ταυτότητες που έχουμε στην Ευρώπη. Θέλω να ξέρουν ποια ήταν η δική μας αντίληψη της ήπιας ισχύω ενδιαφερόντουσαν να ξέρουν πώς αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα συμφιλίωσης. Πέραν αυτών των παραδοσιακών λοιπόν θεμάτων της ανταλλαγής απόψεων και τα λοιπά, θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει την πολιτική κουλτούρα και να τονώσει το ενδιαφέρον για τη δική μας κουλτούρα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ έχει μεγάλες δυνατότητες σε ό,τι αφορά το να μπορέσει να ενισχύσει τις σχέσεις μας με τους εταίρους μας μέσω των εκθέσεών μας και μέσω των ε, υπηρεσιών υποστήριξης των βουλευτών, της κοινοβουλευτικής υπηρεσίας, τεκμηρίωσης κτλ. Έχουμε λοιπόν όλα αυτά τα εργαλεία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να ενθαρρύνουμε περισσότερο την ενίσχυση της πολιτιστικής συνεργασίας. Ευχαριστώ. Vital. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να καλωσορίσω το γεγονό ότι σήμερα συζητάμε τα θέματα πολιτισμού. Γιατί στο μορφότυπο στον οποίο θα συζητάμε τα πράγματα αυτά σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα ήταν ακόμα καλύτερα να είχαμε και λίγη θέρμανση στην αίθουσα, να σα πω την αλήθεια. Τι να κάνουμε όμω. Ο πολιτισμό δεν θα έχει πολύ θέρμανση σήμερα, τι να γίνει. Και χαιρόμαστε που θα θέλαμε μάλλον να υπάρχει και πιο πολύ ενδιαφέρον, όπως είπε ο κ. Πέταρλα, ίσως αυτό να ζέστανε και την αίθουσα. Νομίζω λοιπόν ότι σε ό,τι αφορά την ανακοίνωση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα με ενδιαφέρε να την δω, γιατί δεν την ε, έχω υπόψη μου κανονικά όταν συζητάμε τέτοια θέματα όπως το σημερινό. Έχουμε και κάτι χειροπιαστό μπροστά μας, κάποιο έγγραφο. Αυτό δεν το έχουμε λοιπόν σήμερα. Γιατί ασφαλώς και συζητάμε και συμφωνούμε με όλους όσους μίλησαν σήμερα και είπαν ότι ο πολιτισμός ε, περιλαμβάνει και ορίζει την ευρωπαϊκή ταυτότητα, δίνει αν θέλετε ένα ειδικό βάρος στην Ευρωπαϊκή μας Ένωση σε ό,τι αφορά και τις διεθνείς σχέσεις. Αυτό προφανώς αποτελεί πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Θα πρέπει να γνωρίζουμε επίσης πώς μπορεί να μεταφραστεί σε συγκεκριμένα μέτρα για να μην είμαστε φαφλατάδες και να μιλάμε μόνο, αλλά να εξασφαλίσουμε ότι πρόκειται για πραγματική ανταλλαγή αξιών και όμορφων στοιχείων. Και εδώ λοιπόν θεωρούμε ότι αντιμετωπίζουμε εμπόδια σε ό,τι αφορά το οργανωτικό επίπεδο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν συζητάμε λοιπόν τον πολιτισμό σημασία έχει ιδιαίτερη και η επικουρικότητα, πιο μεγάλη σημασία από ό,τι σε άλλους τομείς. Και αυτό γιατί εδώ πρόκειται για έναν τομέα όπου δημιουργούνται πολλά εμπόδια. Αναφερθήκε το Ινστιτούτο Γκέτε και άλλα τέτοια ιδρύματα μεγάλων ευρωπαϊκών κρατών. Αλλά αυτό που θεωρώ ότι αποτελεί μεγάλο πρόβλημα είναι το εξή ο πολιτισμικός κλάδος σε πολλά κράτη-μέλη δεν διοργανώνεται με τέτοιο τρόπο και η μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών δεν διαθέτει αντίστοιχα τέτοια ιδρύματα πρόθεση του πολιτισμού. Ίσως λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλά θα έκανε να λάβει μια πρωτοβουλία για να προωθήσει τέτοια ιδρύματα. Θα πρέπει να οργανωθούμε. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι η ευρωπαϊκή εκπροσώπηση σε ό,τι αφορά θέματα πολιτισμικά θα διακατέχεται και από μια ισότητα και μια σωστή εκπροσώπηση των κρατών μελών. Και αυτή η ιδέα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μια υπερδύναμη Πρέπει να σας πω ότι ο πολιτισμός θα μείνει κενός νοήματος αν δεν χρησιμοποιήσουμε αυτή τη ε, δύναμη. Ε, σε ό,τι αφορά τον διαπολιτισμικό διάλογο, όλε οι απόπειρε έχουν αποτύχει στο παρελθόν. Θα πρέπει λοιπόν να καταβάλουμε πιο πολλέ προσπάθειες προ την κατεύθυνση αυτή στο μέλλον και να υπάρχει και μεγαλύτερη ειλικρίνεια, να κατανοήσουμε άλλε θρησκείε, άλλου πολιτισμού. Εδώ δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε δραστηριοποιηθεί επαρκώ. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε λοιπόν τι ε, συνέπειε σήμερα αναγκαστικά τι αντιμετωπίζουμε και είναι και πάρα πολύ σημαντικέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει η Πρόεδρο. Και θα ακούσουμε και τον τελευταίο, μάλλον ακούσαμε τον τελευταίο συνάδελφο που είχε ζητήσει το λόγο, να δώσω το λόγο για απαντήσει τώρα, γιατί ακούσαμε και συγκεκριμένα ερωτήματα. Στον κύριο Μαράνη πρώτα. Giving you a general perspective να σας δώσω μια γενική επισκόπηση τώρα για τα ερωτήματα τα οποία τέθηκαν. Βέβαια τα ερωτήματα έχουν αντιμετωπίσει πάρα πολλά ζητήματα τα οποία πράγματι διαλαμβάνονται και στην ανακοίνωση της Κομισιόν. Οι πολιτιστικές διαδρομές είναι κάτι το οποίο το έχουμε υπογραμμίσει ως ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την πολιτιστική μας πολιτική. Όταν αυτές οι διαδρομές βέβαια βρίσκονται μέσα στην Ευρώπη, αυτό δεν έχει να κάνει με την εξωτερική μας πολιτική. Υπάρχει όμως τρόπος να διευρύνουμε, να επεκτείνουμε αυτές τις διαδρομές και εκτός του ευρωπαϊκού εδάφους και ορισμένοι, ορισμένες από αυτές τις διαδρομές ήδη λαμβάνουν υπόψη αυτό το στοιχείο, ιδίως στα Βαλκάνια. Συνεργαζόμαστε μαζί με το Συμβούλιο της Ευρώπης για το εγχείρημα αυτό και εξετάσουμε και δυνατότητα συνεργασία σε ορισμένα σχέδια μαζί με την UNESCO για να αναπτύξουμε τέτοιου είδους προγράμματα τα οποία περιλαμβάνουν τις πολιτιστικές διαδρομές. Γνωρίζουμε βέβαια ότι μπορούν να αποτελέσουν μια ευκαιρία διαλόγου, διαπολιτιστικού διαλόγου και επίσης ανάπτυξης για να προωθήσουν και τη γνώση των γλωσσών, την πολυγλωσσία, την καλύτερη κατανόηση σε περιοχές που έχουν περάσει ταραχώδεις καιρούς στο παρελθόν. Επίσης και τα επιστημονικά θέματα λαμβάνονται υπόψη στην ε, ανακοίνωσή μας. Είναι δυστυχώς αδύνατο να επεκταθούμε υπερβολικά στον τομέα αυτό γιατί παραμένει η ανακοίνωσή μας, μια ανακοίνωση για τα πολιτιστικά θέματα, ακόμα και αν αντιληφθούμε την κουλτούρα με την ευρύτερη δυνατή έννοια, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις πτυχές της υπήρξαν πολλές ε, προτάσεις και συστάσεις που περιλαμβάνονται στις ε, παρεμβάσεις σας. Η ιδέα των κλόουν χωρίς σύνορα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα. Τα τσίρκα είναι ένα στοιχείο πολιτιστικού πλούτου που πρέπει να το διατηρήσουμε και να το προωθήσουμε. Και η ανακοίνωση αυτή μας δίνει και δυνατότητες να το πετύχουμε αυτό. Πρέπει να πω και πάλι ότι από γενική έποψη, γιατί για τις λεπτομέρειες και τα πιο δύσκολα θέματα εγώ θα κάνω πάσα το θέμα αυτό στην Κομισιόν, πρέπει να πω ότι η ανακοίνωση αυτή δίνει δυνατότητες να έχουμε πρόσβαση σε, όλα τα, σε όλες τις πτυχές του πολιτισμού. Εξαρτάται βέβαια από τη θέλησή μας και την κατεύθυνση που θα επιλέξουμε και που θα επιλέξουν τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφωνώ. Για τις καιρικέ συνθήκες που επικρατούν σε αυτή την αίθουσα, νομίζω ότι ο συνάδελφός μας από την Σλοβενία είχε δίκιο λέγοντας ότι επικρατεί ψύχος εδώ. Αλλά είναι γεγονός ότι ο πολιτισμός είναι κάτι, ένα δυναμικό το οποίο δεν έχουμε εκμεταλλευτεί στην Αφρική και εκεί έχουμε να διαδραματίσουμε ένα ιδιαίτερο ρόλο Όπως είπε η κυρία Μοκερίνη, μπορούμε λοιπόν να προσφέρουμε την εμπειρία μας και το παράδειγμά μας. Όχι για να τους διδάξουμε, αλλά για να δείξουμε ποιος είναι ο δρόμος που ακολουθήσαμε, ίσως δεν είναι ο βέλτιστος, αλλά έχει αποδώσει καρπούς και έχει εδρεωθεί με το χρόνο η ήπια ισχύ και η δυνατότητα συμφιλίωση και η ειρήνευση είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε μαζί με τα θέματα της πολιτικής κουλτούρας. Εκεί έχουμε λοιπόν κάποια θετικά παραδείγματα να δείξουμε σε άλλες χώρες. Και τώρα σε ό,τι αφορά την περίπτωση του Euronews, αυτό δεν είναι δικός μας τομέας δράσεις και αρμοδιότητες, εδώ υπάρχουν και κάποιοι που είναι πιο αρμόδιοι σε την αίθουσα για να αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Κομισιόν για να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Ο κ. Σαντιέρη έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Τιέκο. Και ο Τιέκο έχει απαντήσει σε πολλά από τα θέματα που ακούσαμε. Αλλά να σας ευχαριστήσω λοιπόν για την υποστήριξή σας και για τις προτάσεις σας, που είναι πολύ χρήσιμες. Δύο πράγματα να αναφέρω. Σε ό,τι αφορά την ενίσχυση του ενδιαφέροντος για το πολιτικό πολιτισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κάνουμε αυτό, το κάνουμε ήδη. Είναι το τμήμα της δημόσιας διπλωματίας της Ευρώπης αυτό. Και στην ανακοίνωση αυτή δεν θέλαμε να, τα να προκαλέσουμε σύγχυση. Γιατί σε ό,τι αφορά τις προσπάθειές μας για τα πολιτισμικά ζητήματα, δεν θέλαμε να δοθει αυτό υπό το πρίσμα της προπαγάνδας. Δεν κάνουμε προπαγάνδα. Η δημόσια διπλωματία έχει να κάνει με την άμεση ε, αναφορά στους πολίτες μιας άλλης χώρας. Δεν έχει να κάνει αυτό με τον πολιτισμό απαραίτητα. Θέλαμε λοιπόν να κάνουμε αυτή τη διάκριση, αλλά ασφαλώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολείται και με τα θέματα δημόσιας διπλωματίας και όλα τα μέσα που περιλαμβάνονται σε αυτή, σε ό,τι αφορά τώρα τα πολιτισμικά ιδρύματα γιατί άκουσα δύο διαφορετικές απόψεις από αυτού. Καταρχάς, ότι κάνουν εξαιρετικό έργο και ότι θα πρέπει να τι ενθαρρύνουμε, να τα ενθαρρύνουμε να κάνουν πιο πολύ ευρωπαϊκό έργο και όχι τόσο πολύ ξεχωριστά για κάθε χώρα, για την Ισπανία, την Ιταλία, την, τον Εμένα Βασίλειο. Να τι ενθαρρύνουμε, να τα ενθαρρύνουμε να δρουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και κάτι άλλο είναι ότι δεν έχουν όλα τα κράτη-μέλη τέτοια ιδρύματα ανεξάρτητα μέσω στη χρηματοδότηση και το καθεξής. Άρα, τι θέλουμε να κάνουμε, θα πρέπει να συνεργαστούμε και να εργαστούμε πιο πολύ με τις ε, μεγαλύτερες οργανώσεις, προκειμένου να αναπτυχθεί μια ευρωπαϊκή προσέγγιση. Μπορούμε να περιμένουμε βέβαια μέχρι να υπάρχουν σωστοί όροι και σωστέ συνθήκε, αλλά αυτό μπορεί να πάρει πάρα πολύ καιρό. Και έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε τη δουλειά. Και έτσι αποφασίσαμε ότι το πιο σωστό θα ήταν να βοηθήσουμε τα ιδρύματα αυτά να συνεργαστούν, γιατί είναι το ότι κάποιες χώρες έχουν μεγαλύτερη παράδοση σε αυτά τα ιδρύματα από ότι άλλες. Για τα άλλα σημεία τώρα. Θεωρώ ότι καλύφθηκαν από τον Διέγκο για την επιστημονική διπλωματία. Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, Ορίζοντα ορίζοντας 2020 διατίθεται σε, όλο, σε όλες τις χώρες και τα πιο σημαντικά επιστημονικά έργα μπορούν να επιτευχθούν μόνο με συνεργασία όλων και υπάρχει και ο διαπολιτισμικός διάλογος, ο οποίος ε, ε, είναι για παράδειγμα το αντικείμενο του Εράσμους Μούντους, υπάρχει και επιστημονικός στόχος και αυτό το τμήμα της επιστημονικής ε, διπλωματία αναφέρεται στην ανακοίνωση, όχι τόσο πολύ στη διεθνή συνεργασία, για παράδειγμα, για την καταπολέμηση του καρκίνου, πάρα πολύ έγκυρο φυσικά επιστημονικό έργο, αλλά εμεί αναφέρουμε πιο πολύ τον γενικότερο στόχο τη πολιτισμική συνεργασία. Για το Euronews τώρα, πολύ φοβάμαι ότι δεν διαθέτω πληροφορίες γιατί δεν είναι πολύ απλά θέμα της δικής μου γενική διεύθυνση. Ναι, είναι για τη γενική διεύθυνση Connect, λέει η Πρόεδρος. Τώρα δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Έχουμε ήδη καθυστερήσει, λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις απαντήσεις και... Μήπω οι εισηγητές θέλουν να πάρουν το λόγο. Ε, Εγώ, στην Πριν ε, τι τελικέ παρατηρήσει του συναδέλφου Μπρόκ, θέλω να πω δύο λόγια, γιατί είμαστε και συνεισηγητέ. Ε, Ευχαριστώ πολύ όλους ε, όσοι ήρθατε και πήρατε και το λόγο. Θέλω να σας καθησυχάσω ότι πολλές ανησυχίες ε, δικές σας είναι και δικές μας. Όπως τα όσα είπε ο συνάδελφος Μίγια ήδη τα έχουμε σκεφτεί γιατί αυτό είναι ένας από τους άξονες ε, που θα πρέπει να ενισχυθούν και για τα Ινστιτούτα Πολιτισμού, για τις χώρες όπου δεν υπάρχει ισορροπία δυνάμεων. Ήδη βλέπουμε μια δυνατότητα, για παράδειγμα, ζητάμε οι αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις τρίτες χώρες να μπορέσουν με αυτά τα focal points που προβλέπονται από τον ε, ανακοίνωση να βοηθήσουν ώστε να στηριχθεί μια μεγαλύτερη ορατότητα και να ενισχυθεί η συνεργασία. ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη παρουσία και σταθερή παρουσία ε, στις τρίτες χώρες. Ε, ισορροπία λοιπόν με μεγάλη αξία και δράση συνεργασίας για την πρόθεση των κοινών αξιών. Και κάτι ακόμα. θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τώρα να, να θέτουμε τις προτεραιότητες, να ορίζουμε τις προτεραιότητες, ε, την τριμερή διάλογο για το πρόγραμμα για το ευρωπαϊκό έτος που θα είναι αφιερωμένο στην πολιτιστική κληρονομιά θα είναι ένα έδαφος ε, όπου θα μπορέσουμε να πειραματιστούμε για συντονισμένη δράση Φέτος ε, είχαμε τα 30 χρόνια του αέρασμου, τα 30 χρόνια των ε, διαφόρων διαδρομών, όπως είπαμε, πολιτιστικών διαδρομών. Ε, δεν υπάρχουν μόνο οι ατομικές υποτροφίες κυκλοφορίας, αλλά υπάρχουν και εταιρικέ σχέσεις με τρίτες χώρες, όπως η δράση για την Ευρωπαϊκή Εταιρική Σχέση και που κάνει πράγματα και στο πολιτιστικό τομέα, αλλά και οι διάφορες εταιρικέ σχέσεις που προωθούνται από τα πανεπιστήμια και τα πολιτιστικά εκπαιδευτικά ιδρύματα με τρίτε χώρε ε, θα πρέπει να υπάρξει πιο καλή οργάνωση από πλευρά τη Ευρώπη και τη Κομισιόν και βεβαίω υπό την αιγίδα τη Ευρωπαϊκή Εξωτερικής πολιτική ε, για χάραξη συγκεκριμένων και στρατηγικών ε, ώστε να υπάρξει μια σωστή διακυβέρνηση όλη αυτή τη διαδικασία, ώστε να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αυτά δίνω το λόγο βεβαίω στον συμπρόεδρο Μπροκ. Σε ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο Μπροκ. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω αν έχετε προτάσεις να μας ε, το φέρετε στη γνώση μας ώστε να γνωρίζουμε αν υπάρχουν και συγκεκριμένες προτάσεις που μπορούμε να διατυπώσουμε για τα θέματα αυτά. ώστε να μπορέσουν ήδη να περιληφθούν ενδεχομένως τα πρώτα προσχέδια της έκθεσης μας για το θέμα αυτό. Στις 22 Μαρτίου θα παρουσιαστεί η έκθεση ενώπιον της Επιτροπής μας και θα έχουμε βέβαια και τους ε, καλεσμένους μας από την Επιτροπή Πολιτισμού, ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε την περαιτέρω δράση μας. Ο στόχος είναι στις 30 Μαΐου να γίνει η τελική ψηφοφορία, ώστε να μπορέσει να έρθει το θέμα στην Ολομέλεια πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Αυτός λοιπόν θα είναι ο στόχος μας, λέει ο Πρόεδρος τον Ιούλιο, αν θέλει ο Θεός, να έρθει στην Ολομέλεια. Νομίζω ότι είναι η πιο εύλογη διαδικασία. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω, κυρία Κώστα, για την πρωτοβουλία <clears throat> διοργάνωσης αυτής της ε, κοινή ε, συνάντησης. Εγώ πιστεύω ότι μόνο χάρη στη βοήθειά σας θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε